Ε, το καλό του λαού τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τους βοηθήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ελπίζουμε η κατάσταση στην Αλβανία να εξομαλυνθεί και κλείνω τη συζήτηση με αυτή την ιδέα και συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα της της διάταξης που είναι η δήλωση της Επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο υποκλοπής κλήσεων στη Βουλγαρία. Και πρώτα θα ήθελα να ζητήσω την Επίτροπο Πίμπαλξ να, λάβει το, το, να το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προστατεύει το εμπιστευτικό των τηλεφωνικών ε, επικοινωνιών και ε, απαγορεύει κάθε είδους επιτήρηση και παρακολούθηση, μυστική παρακολούθηση του περιεχομένου των κλήσεων. Πέρα από τη νομική απέτηση ε, κατόπιν ε, νομικής κάλυψης για κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητε όπως εμπορικές συναλλαγές, επίσης απαγορεύεται τέτοιου είδους υποκλοπή και σε περίπτωση ε, άρσης τη απαγόρευση αυτής υπόκειται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συνθήκες για τέτοια κατεξαίρεση ε, άδεια υποκλοπή πρέπει να παρέχονται από το δίκαιο και πρέπει να είναι ανάλογες ε, σε μια καταναλογία σε μια δημοκρατική κοινωνία για να διασφαλίζονται τα δημόσια συμφέρον, όπως να υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας ή καταπολέμηση εγκλημάτων οι γενικέ αρχέ και, του... και, οι γενικέ αρχέ του κοινωνικού δικαίου θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βουλγαρική νομοθεσία φαίνεται να συμμορφώνεται προ απαιτήσει αυτέ. Ε, ο νόμος ό,τι αφορά τις ειδικέ ανακριτικές και ε, μεθόδους και μέσα και ο νόμος περί ε, υποκλοπής κλήσεων προβλέπει και σχετική ε, εισαγγελική εξιοδότηση για την πρόσβαση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και εξασφαλίζει πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διακυβευόμενο εδώ είναι ότι η επιβολή και εφαρμογή αυτών των νομικών υποχρεώσεων είναι αρμοδιότητα βεβαίω και ευθύνη των βουλγαρικών αρχών που θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νομικές και διαδικαστικές ε, εγγύησεις θα πρέπει να εφαρμόζονται και να γίνονται σεβαστές εφόσον γίνεται, χρία, γίνεται χρήση αυτών των έκτακτων ε, μεθόδων παρακολούθησης και ανάκρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά ακριβώς από τις βουλγαρικές αρχές να εφαρμόζουν σωστά τις αρχές αυτές, συμμορφούμενοι προς τους κανόνες δικαίου στην εφαρμογή και του σχετικού κοινοτικού δικαίου. Κατανοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι βουλγαρικές αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να ελέγξουν την νομιμότητα της ανάπτυξης τέτοιων ε, ειδικών και έκτακτων διερευνητικών μέσων και προκειμένου να ε, να δουν κατά πόσον η δημοσίευση τέτοιων προσωπικών δεδομένων έχουν προκύψει από κατάχρηση τέτοιων ε, διερευνητικών μεθόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει ιδιαίτερες καταγγελίες και παράπονα ε, ή καταγγελία σε ό,τι αφορά την υποκολοπή κλήσεων ή την χρήση αφαίρετη χρήση τέτοιων στοιχείων. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από το συνεχή την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, και τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων Καταχάσω ο κύριος Πουσοτήλ για τρία λεπτά εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την... Ε, το συζητήσαμε το θέμα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, πρωτού τεθεί εδώ. Το το θέμα το οποίο ε, εδώ πέρα είναι η νομότυπη, η χρήση ε, τέτοιων έκτακτων αθλητικών μεθόδων. Αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι η Βουλγαρία ε, είναι σοβαρή και αντιμετωπίζει την πρόκληση της καταπολέμησης της διαφθοράς και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, όπως ζητήσαμε να το κάνει. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία από τον νόμο ε, εφαρμόζονται με νόμιμο τρόπο και προσδοκούμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Ο νόμο προβλέπει ότι η υποκλοπή κλήσεων μπορεί να ζητηθεί και να παραγγελθεί μόνο από του αγγελείς ή από την αστυνομία και την ε, διεθνή υπηρεσία ασφάλεια, εάν υποψιάζονται το ε, λόγο άτομο εμπλέκεται σε ποινική δραστηριότητα, σε εγκληματική δραστηριότητα και μετά από ξεδότηση του δικαστικού σώματος. Έτσι λοιπόν, ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο ορίζει ρητά ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το μοναδικό σκοπό της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος ή για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους λόγους οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς από τον νόμο. Υπάρχει επίσης και ε, θεσπισμένος κοινοβουλευτικό έλεγχο τη όλη διαδικασία. Άρα είναι σαφέ ότι υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα, τον σεβασμό του απορρίτου και τη ιδιωτικότητα των πολιτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένω, δεν βλέπω να υπάρχει ε, παράβαση του νόμου εδώ πέρα. Επομένω, το να πλήξουμε αυτή τη στιγμή το δίκαιο αυτή τη στιγμή θα είναι ουσιαστικά μια πλήξη της πολύ θεμητής προσπάθειας ενός κράτους μέλους να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Κάποια τέτοιου είδους επίθεση πλήττει την Βουλγαρία, γιατί αυτή η μάχη είναι ύψης για τη χώρα εν ώψη της συνεργασίας και των μηχανισμών επαλήθευσης που διαθέτει και εν ώψη της μελλοντικής ένταξής της στην ε, στη ζώνη Σέγγεν. Η μόνη πιθανή επεξήγηση για την όλη συζήτηση είναι ότι υποκινείται από πολιτικά κίνητρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, ήμουν έτοιμο να χτυπήσω το σφυράκι μου, αλλά τηρήσατε το χρόνο. Επόμενο ο μιλητή, ο κύριο Βόποτα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς ε, που ήταν υπέρ της ένταξης Βουλγαρίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που έγινε μέλος. Αλλά μετά απογοητεύομαι από κάποια από τα μέτρα που λαμβάνει η βουλγαρική κυβέρνηση. Ναι, υποστηρίζουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι κάτι το πολύ σημαντικό και υποστηρίζουμε πλήρως αυτό το οποίο είπε ο Επίτροπος, πως ε, βεβαίως Πρέπει να υπάρχουν νόμοι στη Βουλγαρία και για τις υποκλοπές. Ο Επίτροπος πολύ προσεκτικά είπε φαίνεται πώς συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είπε σαφώς πως πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα των μέτρων. Είναι αναλογικό ξαφνικά μέσα σε τρία χρόνια να περάσουμε από 6.000 υποκλοπές το 2008 σε 16.000 το 2010. Είναι αναλογικό και δίκαιο μόνο 2% των υποκλοπών να καταλήγει στα δικαστήρια και χρησιμοποιείται για το 1% των, καταδίκαιων, των καταδικών. Είναι δίκαιο και αναλογικό να περνάνε διαδικασίες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί δεν πάνε όλα στα δικαστήρια. Γιατί περνάει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών με αυτά τα στοιχεία και Θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να εξετάσει τη διαδικασία ε, εκεί πέρα και των υπολείπων δεδομένων. Και αυτό ακούστηκε και στην Σόφια και στη ε, ΜΜΕ της Βουλγαρίας πως υπάρχουν ε, σοβαρές αμφιβολίες για το εάν μπορεί να προστατεύσει πληροφορίες. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ήδη. Αναφέρατε τη Σέγγεν, ναι θέλουμε τα σύνορα να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αλλά αν δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, θα εκπλαγούμε για το ότι κάποιοι στην Ευρώπη είναι επικριτικοί όσον αφορά αυτή τη διεύρυνση. Πρέπει λοιπόν ο Επίτροπος να, ζητήσει από τη βουλγαρική κυβέρνηση να σταματήσει αυτή τη λανθασμένη εφαρμογή του νόμου, να περάσει σε πολύ δηλαδή περιοριστικές πρακτικές όσον αφορά τις υποκλοπές, να είναι ανοιχτή, διάφανη, δίκαιη και να σταματήσει την παραβίαση τουλάχιστον του πνεύματος του ευρωπαϊκού δικαίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στογιάνοφ έχει σηκώσει την μπλε κάρτα και θέλει να απευθύνει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Αναφερθήκατε σήμερα σε στοιχεία του 2008 και 2010. Αντίστοιχα, από ποια πηγή προέρχονται και πείτε μου, πιστεύετε πως τα στοιχεία αυτά είναι ορθά. Είπατε πως μόνο το 1 με 2% των του προϊόντος των παρακολουθήσεων έχει χρησιμοποιηθεί σε ε, δικαστήρια, αλλά τα στοιχεία που έχουμε εμείς στην Βουλγαρία διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά τα οποία εσείς παρουσιάσατε. Για τα άτομα δηλαδή που ήταν τα αντικείμενα κάποιας ε, τέτοιου είδους παρακολούθησης. Δηλαδή έχουμε 40% ε, του περιεχομένου αυτού που έχουν πάει στα δικαστήρια και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που είπατε εσείς. Έχουμε διαφορετικούς αριθμούς, αλλά από βουλγαρικές πηγές. Ίσως όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει ποια είναι τα σωστά. Από τις διάφορες πηγές που έχω εγώ στη Βουλγαρία, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό το οποίο παραδίδεται στους εισαγγελείς και μετά είναι και πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτού του μικρού ποσοστού που οδηγεί σε ε, καταδικαστικές αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές από, προέρχονται από πολλές πηγές. Έχουμε και μια κοινοβουλευτική έκθεση από τη Βουλγαρία. Πιστεύω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το εξετάσει. Γιατί έχουμε τέτοιου είδους σκάνδαλο στη Βουλγαρία. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους σκάνδαλα. Ε, νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να εξετάσουμε το για ποιο λόγο συνέβη. Κύριε Σόντα, δέχεστε αυτή την μπλε κάρτα που έχει σηκώσει και ο κύριος Γιάννοφ και πάλι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να κάνω λοιπόν μια σύντομη ερώτηση. Μιλάτε για έρευνες που διεξάγουν ε, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, αυτό αληθεύει. Όμως αυτό έγινε κατόπιν απόφασης ε, ε, των σοσιαλιστών. Οι σοσιαλιστές άλλωστε που ανήκουν στη δική σας ομάδα. Look, <laughs> Mr. Κύριε Στογιάνοφ, για μένα δεν έχει να κάνει με κομματική ε, τοποθέτηση έχει να κάνει με το σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου και των κανόνων του δικαίου. Όποιο αποφάσισε να μεταβερθούν αυτέ οι αρμοδιότητε στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι κάτι που δεν με αφορά. Και δεύτερον, είναι η χρήση που γίνεται αυτού του εργαλείου που ε, θα έπρεπε να μας ασχολεί. Μπορεί να χρησιμοποιείται με πολύ ανοιχτό τρόπο και σε πολύ περιορισμένο αριθμό ή το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται πιο διαδεδομένα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε τι συμβαίνει με τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται και παραμένουν μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί εκεί πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος του να ε, συλλέγονται ε, τα στοιχεία αυτά, να διατηρούνται και κατόπιν να γίνεται και κατάχρηση αυτών. Νομίζω πως τέτοιου είδους κατάχρηση θα πρέπει να μας απασχολεί και θα πρέπει εδώ να δράσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Ντάιανα δύο δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ για την πολύ προσεκτική δήλωσή σας. Όσοι με γνωρίζουν στο Κοινοβούλιο και ξέρουν ότι είμαι εδώ 12 χρόνια, ξέρουν ότι έχω παρέμβει, παρεμβαίνω σε τέτοιες με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα και προσοχή. Αλλά ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου αυτού πριν από ένα χρόνο, ήμουν προσκεκλημένη να επισκεφθώ τη Βουλγαρία για να μιλήσω, να παρουσιάσω το σχέδιο στο Στόκχολμ για τη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα αυτό κινήθηκε από την, μετακινήθηκε από το να δίνει την έμφαση στην ασφάλεια στο να δίνει έμφαση στο θέμα της δικαιοσύνης και όλοι προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα αυτά τα δύο. Θυμάμαι από την επίσκεψή μου στην Βουλγαρία το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των Βουλγάρων δικαστών σε, στην δουλειά μας και σε αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε σε κοινοτικό επίπεδο. Εξυπλάγει όμω την περασμένη εβδομάδα όταν, έλαβα μια, όταν είχα μια επίσκεψη στο γραφείο μου στι Βρυξέλλε, όπου μιλούσαν για τη Βουλγαρία, λέγοντα ότι άνθρωποι δέχονταν ε, νύχτα επισκέψεις ε, από άτομα μυστική υπηρεσία κατοίκων. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και να το κατανοήσω και με μεγάλη δυσκολία το ξεστομίζω εδώ. Αυτό λεχθέντες, λοιπόν μου φαίνεται, όπως είπε ήδη ο κ. Βόποντα, ότι η ενισχύει νομοθεσία σε σχέση με τις υποκλοπές κλήσεων, ας τα πούμε όσο έχουν τα πράγματα από το όνομά τους, φαίνεται να είναι σωστή. Όμως ε, υπήρχε μια, αν θέλετε, επίσημη, επίσημος έλεγχος από έναν εξάρτητο σώμα και τώρα από μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτό όμω φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια ε, περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται να υπάρχει ένας, μια αύξηση στον αριθμό των υποκλοπών και φαίνεται, και υπογραμμίζω αυτό το φαίνεται, ότι υπάρχει μια πολύ ευκολότερη και γρηγορότερη εξουσιοδότηση και αδειοδότηση αυτής της δυνατότητας από το δικαστικό σώμα. Ένα συνδεδεμένο θέμα το οποίο θέλω να απτύξω ε, συνδέεται με μια πρωτοβουλία πολιτών που έχει αναπτυχθεί. Φαίνεται ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι υφίστανται πίεση για να αποσύρουν κάποιες υπογραφίες, υπογραφές. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και προσεκτικά το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ευχαριστώ τώρα για την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, ο κύριος Πάσκα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χρησιμοποίηση ειδικών μέσων για την παρακολούθηση είναι παντού ένα ευαίσθητο ζήτημα. Παντού το κράτος μέλος, ε, το κράτος χρησιμοποιεί ε, αυτά τα μέσα και για, την και για το οργανωμένο έγκλημα αλλά μια φορά και για την ε, αντιπολίτευση αλλά στην Βουλγαρία βλέπετε πως έχουν αποθηκευτεί κάποια δεδομένα τα οποία μετά εμφανίζονται από υποκλοπές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό δεν είναι φυσιολογικό ο δε αρμόδιος υπουργός είπε πως γίνονταν κάποιες υποκλοπές για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά δεν συμβαίνει συχνά. Ο Πρωθυπουργό να έχει τέτοια εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του, έτσι ώστε να βάζει να τους παρακολουθούν. Ε, αυτό δεν είναι θέμα εγκληματικότητας. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη η βουλγαρική κατάσταση και πρέπει να βοηθήσουμε τους βουλγαρούς φίλους μας για να εκπληρώσουν ε, τις ε, υποχρεώσεις τους για την βελτίωση νομοθεσίας. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συγχωρείτε, δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο αν έχετε μπλε κάρτα, γιατί όλοι θέλουν να πούν κάτι άλλο και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Οπότε σας παρακαλώ να μιλήσετε όταν έρθει η σειρά σας. Τώρα για τους μεγεγραμμένους, ο κύριος Στογιάννοφ για μισή λεπτό. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα ερτό στη Βουλγαρία και που υλοποιείται ε, εδώ πέρα σήμερα. Θα λέγαμε ελεύθερα ότι βάλαν το λύκο να φυλάει τα έρμα. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι επισήλθε ο νόμος για να καταπολεχθεί η μαφία και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα έχω ξυλοκοπηθεί και εγώ στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας, μιας πορείας διαμαρτυρίας. Τώρα βλέπουμε λύκους με δωρά προβάτου, όντας και και θεράποντες της όλης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος η, η αστυνομία χτυπούσε τους ειρηνικούς διαδηλωτέ, ενώ τώρα διαμαρτύρονται για τις υποκλοπές. Κατά τη διάρκεια του δικού καθεστώτος ε, εξοκοπήθηκε μέχρι θανάτου αρνητής, ενώ τώρα παραπονιέστε για ε, θέματα παρα, για, για θέματα περιστολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άρση ελευθεροτυπίας. Προσπαθείτε τώρα να χρησιμοποιείτε την όλη συζήτηση για να αποφύγετε και να αποτρέψετε την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν και να ρίξετε τα δικά σας, να τα δικά σας και τα εγκλήματα σε άλλους. Οι ψηφοφόροι δεν είναι τυφλοί. Έχετε πέσει στα τάρταρα και καμία βία δεν πρόκειται να αλλάξει τα γεγονότα αυτά. Oh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τις ε, πολιτικές ομάδες, οι μεμονωμένοι αγορητές. Πρώτος, πρώτη η Μαρία Νεντέλτσεβα. Τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω πως οι συζητήσεις αυτές που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντα αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τα θέματα αυτά. Σήμερα διαπιστώνουμε με ποιο τρόπο η ευρωπαϊκή σκηνή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει κανείς διεφθαρμένους πολιτικούς σκοπούς σε ένα εθνικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε την ευρωπαϊκή ατζέντα να την αντικαταστήσουμε μια εθνική. Και δεν θα έπρεπε αυτό να θεωρηθεί μια εθνικά υπεύθυνη θέση, γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες εξέλεξαν τους ευρωβουλευτές τους οι βουλγαλοί πολίτες και δεν νομίζω πως θα ικανοποιηθούν από τα όσα ακούγονται εδώ βεβαίω, τα συνταγματικά δικαιώματα θα πρέπει να τηρηθούν όμως υπάρχουν και όρια και πέρα από τα όρια αυτά νομίζω πως ε, αν αμφισβητήσιμες ομάδες και αμφισβητούμενα συμφέροντα που προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα θα καταφέρουν τελικά να επιβάλλουν κάποιες διεφθαρμένες πρακτικές και να κακολογήσουν τη Βουλγαρία στα μάτια του κόσμου. Ακούστηκαν κάποιοι υπενιγμοί πως ο αριθμός των υποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων έχει διπλασιαστεί. Τα επίσημα στοιχεία διαφέρουν, αλλά δεν θα σας φέρω αντίρρηση εδώ, θα σας ρωτήσω το εξής. Από πότε ο αριθμός αυτών των υποθέσεων έχει γίνει τόσο σημαντικός ποιοι έδωσαν ανοιχτή πρόσβαση στους πολίτες στον αριθμό αυτών των υποθέσεων, ποιοι επέφεραν τη διαφάνεια εδώ, η δική μας κυβέρνηση και είχαμε αυτή την ε, η αυτόνομη ανεξάρτητη επιτροπή η οποία υποτίθεται παρακολουθούσε την κατάσταση. Αλλά αυτό ποτέ δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Η Βουλγαρία έχει κοινοβουλευτικό, ε, είναι μια δημοκρατία με κοινοβουλευτικό πολίτευμα και ακριβώς γι' αυτό η παρακολούθηση των μυστικών υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχουν όλες οι πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται ε, στη δική μας Βουλή. Βλέπετε λοιπόν πως η βουλγαρική νομοθεσία εξασφαλίζει τα εχέγγυα για την νόμιμη χρήση αυτών των ε, ερευνητικών δυνατοτήτων. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να χτίσει κανείς από το τίποτα κάτι θετικό. Το πιο δύσκολο όμως είναι να διαπιστώνει κανείς πως οι εκπρόσωποι της Βουλγαρίας εδώ προωθούν συμφέροντα πολύ διαφορετικά από τα οποία θα έπρεπε να υποστηρίζουν γιατί άλλος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος μας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω στον επόμενο ομιλητή ε, το λόγο που είναι ο κύριος Μωράης. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. uncomfortable. Κύριε είναι πάντα δύσκολο να εξετάζουμε την εσωτερική κατάσταση σε οποιοδήποτε κράτου μέλους. Οπότε στο πνεύμα της κυρίας Βόλης θα έλεγα και εγώ πως και η δική μου κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ερευνήθηκε για το τι έκανε με τις συλλήψεις και παραδόσεις ανθρώπων στους Αμερικανούς για να βασανιστούν. Αυτό ήταν άβολο και για τη δική μου κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά συμμετείχα ενεργά σε αυτή την έρευνα. Γιατί έπρεπε να γίνει πανευρωπαϊκά. Γιατί λοιπόν και γιατί συζητάμε σήμερα τα εσωτερικά των υποκλοπών της Βουλγαρίας. Όχι λόγω της Βουλγαρίας, αλλά γιατί είμαστε μια κοινότητα αξιών. Ως μια κοινότητα αξιών, τα ζητήματα τα οποία έθιξε ο κ. Επίτροπος αναφέρω πώς πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω εξαίρεση η υποκλοπή. Ε, δεν είμαι φοβερός νομικός όπως η κυρία Γουάλης, αλλά ως νομικός ξέρω πως πρέπει να χρησιμοποιείται πράγματι κατ' εξαίρεση. Η υποκλοπή, αν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ακατάλληλο και δυσανάλογο, αντί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στη Βουλγαρία και άλλο, γίνεται όπλο του κράτους. Και δεν έχει σημασία ποιο πολιτικό κόμμα το ξεκίνησε αυτό. Το να περάσουμε από την επίθεση κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε μια δυσανάλογη χρήση αυτού του μέσου είναι κάτι το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά μόνο τη Βουλγαρία. Σήμερα είναι η Βουλγαρία, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη χώρα. Όσον αφορά τις πηγές και τους αριθμούς, θα ε, Ρώτουσα τους συναδέλφους, λέει κάποιος πως ε, μία λανθασμένη ή δυσανάλογη χρήση δεν έλαβε χώρα. Εάν θέλετε να αμφισβητήσετε τους αριθμούς του, κυρία, του κυρίου Σφόμποντα, αμφισβητεί κανείς την δυσανάλογη χρήση υποκλοπών. Κοίταξα πολλές πηγές πριν μιλήσω σήμερα γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τέτοια ζητήματα και δεν είδα κανέναν πουθενά στην συζήτηση να λέει πως δεν ε, υπήρξε δυσανάλογη χρήση. Γι' αυτό η Κομισιόν πρέπει να το ερευνήσει. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μα συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας ε, διακόψω. Είμαστε κατά των υποκλαπών να το χρησιμοποιούνται παράνομα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που καταπολεμούν τη μαφία και τελευταία έχει χρησιμοποιηθεί όμως και από τον εγκληματία κύριο Μπελουσκόνη για εγκλήματα που δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί, για ε, προαγωγή ανηλίκων. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι τελείω διαφορετική στη Βουλγαρία, γιατί η βουλγαρική κυβέρνηση φαίνεται ότι χρησιμοποιεί το μέσον αυτό των υποκλοπών για να ποινικοποιήσει την αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντα τον διάχυτο φόβο και αποπειρώμενη να ταυτίσει την αντιπολίτευση με κοινού εγκληματίε που θα του επιτρέπει να δράσουν χωρί κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να είναι κράτο αστυνομικό. Μια τέτοια κατάσταση επιδεινώνει ε, την κοινωνική κατάσταση και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, με πολύ ιδιαίτερη προσοχή να παρακολουθούν την κατάσταση στην Βουλγαρία για να περιοριστούν το, να περισσοθούν οι βλάβες που απειλεί να, απειλεί επιφέρει αυτή η στάση της ευρωπαϊκής, της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράσερ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, παρακολούθησα τη συζήτηση αυτή και την προηγούμενη συζήτηση για την Αλβαρία. Ποια, οποία διαφορά Εκεί πέρα διακομματικά προσπαθούμε να βρούμε το σωστό τόνο και εδώ πέρα ακούμε κατηγορίες αναπόδεικτες. Στόχος που από τη μία είναι να καθίσουν σε ένα τραπέζι τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά από την άλλη είναι να μην υπάρξει συμπαιχνία των δύο μεγάλων κομμάτων. Από τη μία η επιθυμία τα κόμματα να βοηθήσουν τον λαό και να συνεργαστούν και εδώ πέρα πάλι δυστυχώς υπάρχει μια λανθασμένη καταδίκη από πλευρά, μία πλευρά του Κοινοβουλίου. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί δεν ακούω ούτε ένα γεγονός αλλά μόνο λέτε μας είπανε κάποιες πηγές, ακούσαμε και τέτοια. Εάν το βλέπετε έτσι, τότε γιατί δεν πάτε εκεί στις αρμόδιες επιτροπές εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Γιατί δεν πάτε στην Επιτροπή Ασφαλείας. Γιατί δεν θέτε ένα ερώτημα προ την Κομισιόν. Όχι. Προκαλείται εδώ πέρα μια ανοιχτή συζήτηση γιατί επιθυμείται αυτή η συζήτηση για πολιτικούς λόγους. Αυτό το απορρίπτουμε. Δεν το θέλουμε. Δεν είναι δυνατόν έτσι να παίζουμε παιχνίδια στην πλάτη του βουλγαρικού λαού και της κυβέρνησης. Εάν υπάρχει κάτι να συζητηθεί, τότε σας παρακαλώ να το κάνετε στην αρμόδια επιτροπή. Είναι αυτονόητο πως πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου, να λειτουργεί η δικαιοσύνη και ειδικά σε ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτό το μέσο να υπάρχει ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος που έκανε αυτή η κυβέρνηση και ξεκίνησε για πρώτη φορά από αυτή την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν όλες οι ομάδες του Κοινοβουλίου και ευχαριστώ την κυρία Μάλμστρομ η οποία δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα πως είναι εσωτερική αυτή η συζήτηση και είπε πως η βουλγαρική κυβέρνηση έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα. Ευχαριστώ. Οποιοςδήποτε ζητάει μπλε ε, κάρτα δεν θα την λάβει. Θα δώσω τον λόγο μόνο σε όσους τον έχουν. Κοιτάξτε, υπήρχε κάποιος εδώ πέρα όρθιος και τραβούσε, και τραβούσε τις υπογραφές και λέει πως είναι από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία. Κινηματογραφούσε, δεν ξέρω. Περίεργο είναι να μπαίνει κάποιος στην αίθουσα, μας κινηματογραφεί όταν μιλάμε. Όχι, όχι, μέσα στην αίθουσα ήταν. Και ε, το παρουσιολόγιο εκεί με τι υπογραφέ Να το δουν οι υπηρεσίε. δεν είναι το να μπαίνουν άσχετοι εδώ μέσα και να κινηματογραφούν. Ε, άμα δεν ξέρει, μην μιλά. θα εμπληθούμε τη κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα λάβουμε τα ανάλογα μέτρα. Λοιπόν, μπλε κάρτα. Θα πάρετε μετά το λόγο. Μπορείτε να αντιδράσετε. Παρακαλώ πολύ. Μην ε, διπλασιάζετε το χρόνο παρεμβάσεών σας. Η κυρία Γιώτοβα, ένα λεπτό. Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο στα θέματα υποκλοπών στη Βουλγαρία, αλλά αφορά και τι πολύ ανησυχητικέ τάσει που παίρνουν η προστασία πολιτικών ελευθεριών και πολιτικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη οι βουλγαρικέ αρχέ πρέπει να επιλύσουν αυτό το ιστορικό πρόβλημα. Αλλά σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, η βουλγαρική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί σωστά. Σωστά λέτε, κύριε Επίτροπε. Το πρόβλημα έγκυται στο θέμα της εφαρμογής του νόμου αυτού. Και γι' αυτό ρωτάμε τον Επίτροπο, τι θα κάνετε ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση του κοινοτικού δικαίου. Ε, δικαίου συγγνώμη. Η ερώτηση αυτή είναι του κ. Στράσερ. Και το πρόγραμμα στο Στοκχόλμη και η Οδηγία 9496 και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διακυβεύεται. Γιατί αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν υποκλοπέ που γίνονται και από γιατρού χωρί νομική νομοποίηση και χωρί τη δυνατότητα ατόμων να υπερασπιστούν του εαυτού του στα δικαστήρια αυτής ο διπλασιασμός τελικά των περιπτώσεων υποκλοπών είναι αντιστρόφως ανάλογος με την επιτυχή ε, εκδίκαση υποθέσεων και αριθμό εκδίκασης υποθέσεων σχετικά στα δικαστήρια. Κύριε Πέτροπε, οι ειδικέ ανακριτικέ και ερευνητικέ μέθοδοι είναι απαραίτητε για την πολέμηση του εγκλήματο και παρακαλούμε πολύ να παρακολουθήσετε πολύ κοντά την παράτυπη εφαρμογή των μεθόδων αυτών στα πλαίσια του μηχανισμού συνεργασίας. Ε, ευχαριστώ, Στάνιμιρ Ήλτσεφ, για δύο λεπτά. Κύριε Ήλτσεφ. ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η χρήση των ειδικών αυτών ε, μέσων έρευνας έχει κλιμακωθεί στη Βουλγαρία, γι' αυτό η κοινή γνώμη ενισχύει. Είναι ο κοινοβουλευτικός φορέας του Κοινοβουλίου που επιτηρεί αυτές τις υποθέσεις που έχει κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις επικριτικές και ζητώ να τις διαβάσετε. Και κατόπιν, ποιο θα είναι το μήνυμα της Κομισιόν προς εκείνους που δεν ξέρουν ποια είναι η λεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Θα, τους, ε, θα καταδικάσει η Κομισιόν όσους χρησιμοποιούν πόρους του κράτους για προσωπικά και πολιτικά συμφέροντα και πόσο αυστηρή θα είναι η Κομισιόν στο να ζητήσει να πληρωθούν κάποια προφανή νομοθετικά και να είναι σαφές πως οι ε, λάθρα αυτές από πληροφορίες ε, δεν έχουν πάει μόνο σε ερευνητικέ ομάδες αλλά και σε πολιτικούς αξιωματούχους. Οι αστυνομικοί φιλτράρουν τις πληροφορίες και δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Η έγκριση ε, για τις ε, υποκλοπές δεν ε, είναι πάντα δικαιολογημένοι. Οι δε βουλγαρικές αρχές ασφαλείας έχουν αναπτύξει περίεργα αντανακλαστικά. Οτιδήποτε κινείται παρακολουθείτε. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι δικαστές και όχι οι πολιτικοί λένε πως είτε το σύστημα έχει λάθος ή πως ε, πρόκειται για μία περίπτωση κοταδισμού. Και βεβαίως ε, αν είναι θέμα σκοταδισμού πρέπει να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή και τις ελευθερίες. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης δεν είναι έκθεμα μουσείου. Έχει στόχο να γίνει η Ευρώπη ένα στόχος ε, ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας και δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κόβατσεφ έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, αυτό που ακούσαμε από τον, Επιτροπό την νομοθεσία στη Βουλγαρία που είναι εφαρμοστέα στην χρήση ειδικών διερευνητικών μεθόδων, ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό δίκαιο. Δεν διαφωνούμε στο ότι κάθε κράτης μέλος θα πρέπει να εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικαστικών ε, δικαιωμάτων. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει προκληθεί σήμερα. Είναι πολύ απλό. Ξεκινά μια προεκλογική εκστρατεία στην Βουλγαρία, προεκλογική περίοδος και μεταφέρονται οι αντιπαλότητες σε, στο θέατρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι να υπάρξει μεγαλύτερο πολιτικό μέρισμα. Είναι δύσκολο όμως να πιστούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τις καλές προθέσεις των ανώτερων, των ηγετών των τριών ε, κομμάτων συνασπισμού, κυβερνητικού συνασπισμού της Βουλγαρίας. Υπήρξαν πολλά περιπτώσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων στο παρελθόν. Κάποιοι δεν περίμεναν να ακούσουν, ε, να πάρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που υπέβαλαν. Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι αυτοί, οι οποίοι έφυγαν από την αίθουσα, καθοδηγούνται στις προθέσεις τους από την ιδέα να πλήξουν στο δυνατόν περισσότερο την βουλγαρική κυβέρνηση. Είμαστε Βούλγαροι εναντίον Βουλγάρων σε αυτή την Ολομέλεια σήμερα, αντί να συνεργαζόμαστε. Η σημερινή κυβέρνηση δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο λόγω των υπολοιμάτων και των σταγονιδίων της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο στόχος εδώ δεν είναι μόνο να αρθεί η αξιοπιστία του κυβερνώντος κόμματος, αλλά να, ε, να τρωθεί η αξιοπιστία όλη τη χώρα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα είναι πονίδιστο και πραγματικά αξιοθρύνητο. Κατά τη διάρκεια των ε, τελευταίων, των πρόσφατων ημερών οι βούλγαροι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση έχουν πραγματικά ζωγραφίσει με τα μελανότερα χρώματα την πολιτική σκηνή στη Βουλγαρία. Ακούσαμε περί σκοταδισμού, περί φτώγιας, περί λοιμού. Όλες αυτές είναι σαφείς πολιτικές απόπειρε να μαυρωθεί η Βουλγαρία. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Δεν υπάρχουν ε, συμβόλαια θανάτου τα κύρια, ε, οι κύρια διάβλοι ε, διαφθοράς έχουν αποκοπεί. Όλα αυτά τα κανάλια που γέμιζαν τους, ε, τις τσέπες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έχουμε δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό επενδυτικό περιβάλλον στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση έχει σταθερή πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο και συμμετέχει σε όλες τις ευρωπαϊκές διαδικασίες σαν αξιόπιστο συνομιλητή. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους παριστάμενου ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές. Πραγματικά σπαταλάμε το χρόνο εξαιτία του ότι βρισκόμαστε προκλογική περίοδο στη Βουλγαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Εντσού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των παράνομων υποκλοπών στη Βουλγαρία είναι εξαιρετικά σοβαρή. Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ε, σημειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, η συζήτηση αυτή θα έπρεπε να είχε αναφερθεί και σε άλλη μια χώρα, την, στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία το 2011 οι υποκλοπές ιδιωτικών συνομιλιών ε, ήταν, εξακολουθούν να είναι δυνατές χωρίς καμία νομική κάλυψη. Ενώ και το Σύνταγμα και η εσωτερική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο απαγορεύει την, ε, απαγορεύει την ε, παρακολούθηση και την παρισύφρηση στην ιδιωτική ζωή χωρίς ειδική εξιοδότηση. Οποιαδήποτε κατάχρηση ε, απαγορε, όπως επίσης ένα θεμελιώδες δικαίωμα που δεν γίνεται σεβαστό, γιατί η κύρια προτιμόμενη μέθοδος των εισαγγελέων είναι η παράνομη παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν συστηματικά τις ε, τηλεφωνικές ε, συνδιαλλαγές ε, των μελών της αντιπολίτευσης. Ζητώ την κατεπίγουσα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τηρηθεί το κράτος δικαίου και η δημοκρατία και στα δύο κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ουρούτσεφ ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πως η βουλγαρική κυβέρνηση ε, επέδειξε αποφασιστικότητα για να στρίψει το οργανωμένο έγκλημα και τη αφορά. Για πρώτη φορά είχαμε απτή πρόοδο. Αυτό επέλεξαν οι Βούλγαροι ψηφοφόροι στις εκλογές του 2009. Όλα τα θεμητά μέσα χρησιμοποιούνται για να ερευνήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Μην είμαστε αφελείς. Το οργανωμένο έγκλημα έχει πολλούς πόρους. που συσσωρεύτηκαν τα έτη της ατιμορρησίας και της αδράνειας και τώρα αντιδρούν. Διασπείρουν έγγραφα τα οποία καθιστούν ανθρώπους αναξιόπιστους και υποκλοπές οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στα ΜΜΕ που διακινούν ε, βιντεοκασέτες, ε, βίντεο και ηχογραφήσεις. Είναι ιστερία πραγματικά. Όλα αυτά ακούγονται ως κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην εξακρίβωση της αλήθειας αλλά στην πραγματικότητα αυτό επιθυμούν οι διάφορες εγκληματικές ε, ομάδες δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών στη Βουλγαρία αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια προσπάθεια να καταστεί η κυβέρνηση αναξιόπιστη και μαζί με αυτό και η θέλησή της να καταπολεμήσει την διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Οι εγκληματίες προσπαθούν να αδρέψουν τους καρπούς των κινήσεών τους εν ώψη των εκλογών που έρχονται. Σκεφτείτε το αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Κάλφιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια προς τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Πόρη προπαγάνδα κυκλοφορεί. Υπάρχει εδώ πέρα ένα μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού. Οι εθνικιστές του ΑΤΑΚΑ έφεραν μια έκθεση στο Κοινοβούλιο που έλεγε πως η κυβέρνηση φιλτράριζε τα στοιχεία πριν τα στείλει στο δικαστήριο. Και η κυβέρνηση αυτή έλεγε πως, ε, η έκθεση έλεγε πως η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία τα οποία καταλήγουν στα ΜΜΕ. Και η έκθεση αυτή έλεγε πως υπήρξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραβιάστηκαν κάποια θεμελιώδη νομοθετήματα και πρέπει να συγκρίνει η Κομισιόν τη βουλγαρική νομοθεσία και την εφαρμογή της σε σύγκριση με το τι γίνεται σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται προπαγάνδα εδώ μέσα, ούτε ιδεολογική μάχη. Πρέπει να ε, δει τα γεγονότα η Κομισιόν και να τα αναλύσει. Ευχαριστώ. Ε, έχει προχωρήσει η ώρα, λυπούμε, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο με βάση την μπλε κάρτα. Οπότε Περνάμε στον κύριο Νέινσκι για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Νέινσκι. Θα ήθελα, μια που είμαι μια από τις τελευταίες ομιλήτριες για τον κατάλογο, να κάνω μια σύνοψη των όσων ακούστηκαν στη συζήτηση σήμερα. Γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει με υποκλοπές, ούτε έχει να κάνει με το κατά πόσο είμαστε υπέρ ή κατά κάποιου συγκεκριμένου υπουργού. Έχει να κάνει με τις αρχές που περτανεύουν στην Ευρώπη και μετά όσο υποστηρίζουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να κάνει με τη δημοκρατία, με, με την ισονομία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν δεν είναι καθαρά εγχώριο θέμα εσωτερικής τάξης. Γιατί νομίζω ότι αυτό που διαπιστώνουμε μετά που γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου είναι πως οι πολίτες όταν χάσουν την πίστη τους στις αρχές χάνουν τα πάντα. Η σημερινή συζήτηση έχει να κάνει με το τι είναι αληθινό και δεν υπάρχει ούτε η μία αλήθεια ούτε χρωματισμένη αλήθεια. Η αλήθεια είναι ενιαία και δεν είναι ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Αυτό που πρέπει να δούμε λοιπόν σήμερα είναι το θέμα της υπευθυνότητας η ευθύνη βέβαια της σημερινής κυβέρνησης, όχι προηγούμενων ή επόμενων κυβερνήσεων, γιατί η κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εξουσία πρέπει να λογοδοτήσει στους πολίτες της. Οι πολίτες αυτοί μπορεί να είναι ψηφοφόροι ή μπορεί να είναι αντιπολιτευόμενοι, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός πεδίου δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να με συγχωρήσετε που ε, δεν σας έδωσα το σωστό όνομα. Εν πάση περιπτώσει θα περάσουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι της διαδικασίας, το Catch the Eye. Έξι έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Ιβάνοβα είναι η πρώτη. Ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μετά τα όσα ακούσαμε, το μόνο που μπορώ να πω είναι πως Για μια φορά ακόμα είδαμε μια λυπηρή προσπάθεια της αντιπολίτευσης Βουλγαρία να δημιουργήσει, να δώσει μια ε, ευρωπαϊκή διάσταση σε ένα θέμα εσωτερικό. και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Βουλγαρίας προσπαθούν να καταστήσουν αναξιόπιστη τη Βουλγαρία στα μάτια των, ευρωπαϊκών, των Ευρωπαίων εταίρων τους. Αυτό διακυβεύεται σήμερα. Θα θυμόμαστε όμως τα σκληρά λόγια που ακούστηκαν σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, εάν δεν μπορεί να είστε επικοδομητικά αυστηροί με την κυβέρνηση ε, της Βουλγαρίας, αν δεν μπορείτε να παράσχετε ε, επικοδομητικές ε, προτάσεις, σας παρακαλώ τουλάχιστον μην παρακολύετε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι επικοδομητικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπίγκανεν έχει το λόγο. Προηγουμένως λόγω μπλε κάρτας δεν σας έδωσα το λόγο, αλλά μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Θα τα πω στα πλαίσια του Catch the Eye, αλλά εγώ είχα ζητήσει μπλε κάρτα για να αντιδράσω, είπε ο κύριο Στράσερ. Τα όσα είπε λοιπόν ο συνάδελφος, με βρίσκουν αντίθετο. Δεν μπορώ να δεχτώ πως δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα τέτοιου είδους μέτρα για να έρευνες αστυνομικές έχουν χρησιμοποιηθεί. Τι έχουμε στην έκθεση, 15.946 εγκρίσεις τέτοιου είδους παρακολουθήσεων και μόνο 1.918 υποθέσεις κατέληξαν στα δικαστήρια. Είναι ελάχιστο το ποσό αυτό. Μιλάμε για σχεδόν 16.000 εγκρίσεις, το οποίο σημαίνει πως 5 με 10% των Βουλγάρων πολιτών ήταν αντικείμενο παρακολούθησης κατά το 2010. Κύριε Στράσερ, αυτά κάνετε στην Αυστρία εσείς. Θα συμφωνούσατε σε τέτοιες πρακτικές στη χώρα σας. Μιλάμε για ελευθερία, για δημοκρατία αλλά για κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παρβάνοβα για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει το εξή. Ξέρετε εσείς στην Επιτροπή πως 27 υποθέσεις που είναι στο δικαστήριο στο Στρασβούργο δικαιώθηκαν οι ενάγοντες οι οποίοι είχαν κατηγορήσει για βαναυσότητα την αστυνομία μας. Μιλάμε για κινήματα πολιτών όπου ζητάνε και πιέζουν τους πολίτες να αποσύρουν υπογραφές από τέτοιου είδους κινήματα και όπου περνάνε ανακρίσεις στα αστυνομικά τμήματα και πολύ συχνά συλλαμβάνονται οι αντίπαλοι της κυβέρνησης. Όσοι θεωρούνται εχθροί της κυβέρνησης θεωρούνται και, και παρουσιάζονται ως εχθροί της κοινωνίας μας. Αυτό κατά τη γνώμη είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Εχθές σε μία επίσημη συνάντηση της ηγεσία μας με την ηγεσία του κόμματος Γκέρμπ πιεστήκαμε να αφαιρέσουμε αυτή την προφορική ερώτηση από την ημερήσια διάταξη. Άρα λοιπόν τι μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, ε, εδραιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στη διαδικασία του KTDI. Σας υπενθυμίζω και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να απευθυνθώ απευθεία σε εσά. Είναι λυπηρό πως ενώ όλοι προσπαθούμε... Ε, δεν έχει νόημα αν, δεν με ακούμε, αν δεν με ακούτε. Προσπαθούμε να κάνουμε πιο ζωντανές συζητήσεις και δεν ε, μας αφήνετε να χρησιμοποιήσουμε την μπλε κάρτα μπορεί να υπάρξει νομίζω μια ποιοτική αναβάθμιση της ε, συζήτησης. Ε, άμα δεν με ακούτε δεν χρειάζεται και να μιλάω κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν έχει νόημα. Ε, υπάρχει ένα συνάδελφος που το έχει πει εδώ πέρα κοινοβούλιο καραόκε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση και δεν μας ακούτε καν δηλαδή, δεν υπάρχουμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μπαλτσίτης. Επί της διαδικασίας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, ήθελα να συμφωνήσω και εγώ πως τα απόψε, πως δεν βλέπετε τις μπλε κάρτες. Και ε, επειδή λένε όλοι πως ε, δεν υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι εδώ πέρα, υπάρχουν αρκετοί αξιοσέβα συνάδελφοι εδώ πέρα που ακούν την συζήτηση. Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου απογοήτευση, κύριε Στράσερ κύριε Στράσερ, πραγματικά δεν ήταν αυτό ε, δείγμα δημοκρατικής ομιλίας ε, και από μια χώρα την οποία σεβόμαστε ως δημοκρατική. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Μπαλτσίτση για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα είναι περίπλοκο. Με βάση λοιπόν τις διαθέσιμες πληροφορίες το πρόβλημα ε, μάλλον υπάρχει. Και συμφωνώ με συναδέλφους που μίλησαν και είπαν πως δεν είναι μόνο βουλγαρικό το ζήτημα. Μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες και όλοι πρέπει να σεβόμαστε όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση σε αυτή την αίθουσα. Εξάλλου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια χάρτα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, και η Βουλγαρία ή η Λιθουανία και όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν αυτή τη χάρτα η οποία περιγράφει σαφώς το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν τα κράτη-μέλη. Το βασικό είναι να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ λοιπόν πως ο κύριος Επίτροπος πρέπει να εξετάσει από κοντά την ε, κατάσταση. Γιατί όπως ε, το βλέπετε και εδώ μέσα η κατάσταση ίσως είναι λίγο τεχνητή και διωγγωμένη. Η κυρία Γιουσμένοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Φυσικό είναι να γίνονται συζητήσεις ε, όταν μιλάμε για σημαντικές ευρωπαϊκές αρχές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό να τα συζητάμε όταν παραβιάζονται ή είναι ευπαθή. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, όλες αυτές οι συζητήσεις ήταν και οι ομιλίες ήταν προς την ίδια κατεύθυνση γιατί εξέφρασαν ανησυχία φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές ε, ευρωβουλευτές ζητήσαμε αυτή τη συζήτηση γιατί ανησυχούμε για το κράτος δικαίου και την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Βουλγαρία. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους ε, ψηφοφόρους μας πως ε, θα είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπίσουμε τις αξίες τους. Είχαμε ανησυχίες από τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ελπίζω λοιπόν αυτές οι κοινέ ανησυχίε να οδηγήσουν σε μια λύση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρινάλδη ζήτησε μπλε κάρτα, οπότε έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι φιλελεύθερο δημοκράτης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ιταλία. Πολύ συχνά στη χώρα μου μαζί με τους συντρόφους του κόμματό μου πολύ συχνά ε, μας, αποκαλούν κομμουνιστές. Απλώς και μόνο γιατί είμαστε ενάντι στην ε, κυβέρνηση που έχει την εξουσία αυτή τη στιγμή στη χώρα μου. Και σε σχέση με αυτά που διαβάζουμε και που προκύπτει, συμβαίνει κάτι στους ε, συναδέλφους είτε σοσιαλιστές είτε φιλελεύθερους στην Βουλγαρία, ορίζονται αν θέλετε και ε, χαρακτηρίζονται σαν εγκληματίε γιατί παραμείνονται τη χώρα του. Δεν μα αρέσει καθόλου αυτή η παρέκκληση γιατί προφανέστατα κάποια τέτοια τάση μπορεί να πάρει και πολύ επικίνδυνες ε, πτυχές και ε, τροπές. Μόλις χθε, μετά από όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και την Ισία, μόλις χθε πήγε ο Υπουργό Εξωτερικών χθε και χαρακτήρισε στη Συρία, στη Δαμασκό, μια χώρα δημοκρατική, η οποία πλήρως ικανοποιεί τις ανάγκες εκδημοκρατισμού και, εκδημοκρατισμού και εξυγχρονισμού των πολιτών τη. Αυτή είναι η κατάσταση, Εμεί πρέπει να το καταγγείλουμε. Αλλά και εσείς, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είστε πραγματικά σε επιφυλακή και να προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα Δίνω τον λόγο στον ε, Επίτροπο, τον κύριο Πίμπαλξ. Εκτός μικροφώνου, Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότυπα μέλη, ήταν πολύ έντονη η συζήτηση, είναι αλήθεια, αλλά θα τονίσω τρία σημεία που πιστεύω ότι είναι θεμελιώδη. Η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική μου χώρα δεν ήταν καθόλου εύκολη. Όταν όμως μια χώρα γίνεται αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι η ιδιότητα αυτή του μέλους της, ε, του να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό λειτουργεί σαν εχέγγυο ε, εφαρμογής και του ευρωπαϊκού δικαίου και σε βασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ειδική νομοθεσία, η οδηγία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών στοιχείων, την προστασία της ιδιωτικότητας, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ μακρά και αξιοσέβαστη θα έλεγα ιστορία ε, παρακολούθησης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε κάποιο κράτος μέλος. Σας ανέφερα ακριβώς πού βρισκόμαστε και πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχετε πλήρη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες της, ότι αν υπάρξει παραβίαση κοινοτικού δικαίου θα δράσει. Εάν όχι, δεν πρόκειται να λάβει δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ασκεί αυτόν τον ρόλο στενή ε, παρακολούθηση και αν απαιτηθεί θα παρέμβει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπερβούμε την εντολή και τις δομές του Ευρωπαϊκού Δικαίου και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θα παραμείνει ε, νομότυπη και θα εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστέψτε με, λέει ο Πρόεδρος, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι ε, ως προερχόμενος από μια πρώην